πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, στο ECR. Δεύτερη ανακοίνωση. Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες ε, θα κάνουμε την εξής αλλαγή Τη ημερήσιας διάταξης για Τετάρτη σήμερα. Ως τελευταίο σημείο προβλεπόντουσαν οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Προστασία των Καταγγελόντων, αποκαλούμενων whistleblowers, θα υπάρξει δήλωση της Κομισιόν επ' αυτού και για την Πέμπτη προβλεπόταν η τελική ψηφοφορία για την έκθεση Χαρνές σχετικά με την εισαγωγή ε, πηγόντων εμπορικών μέτρων για την ε, Τινησία. Ε, αυτό θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης. Αντιρρήσεις παρακαλώ, από ό,τι βλέπω όχι. Ελπίζω να εγκρίνατε αυτές τις αλλαγές της ημερήσιας διάταξης και άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται για προφορική τροπολογία. Είναι μία πρόταση να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Συνάδελφοι, βλέπω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες κατεγράφησαν που σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε στις προτινόμενες αλλαγές τη μερικής διάταξη. Σας ζητώ λοιπόν, ποιος είναι, σας ρωτώ, ποιος είναι υπέρ των προτινόμενων αλλαγών στη ημερήσια διάταξη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται οι αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ.